Είναι μια συζήτηση αυτή που δεν υπάρχει κατσιάι, δηλαδή δεν ζητάτε το λόγο, ε, ούτε γαλάζιες κάρτες έχουμε και μόλις 40 λεπτά για τη συζήτηση. Θα μιλήσει ο Αντιπρόεδρος Εύκοβης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μετά εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων και θα σας παρακαλέσω όλους όσο γίνεται να προσαρμόσετε και να τηρήσετε το χρόνο σας γιατί δεν θα πρέπει ε, να καθυστερήσει η τελετή για το βραβείο Ζαχάροφ. Εξ ονόμα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το λόγο έχει ο αντιπρόεδρο κ. Σεύκοβιτ. Μάρου, έχει το λόγο. Thank you very much, uh, Mr. President, honorable members. Πρόεδρε, κύριε Βουλευτέ, με μεγάλη μου ικανοποίηση να σα παρουσιάσω το ε, πρόγραμμα εργασία του 2014. Πρόκειται για ένα συνδυασμό εντατικού πολιτικού διαλόγου μεταξύ των θεσμικών οργάνων, Οπότε προσπαθούμε να βασιστούμε στη συζήτηση για την κατάσταση Ευρωπαϊκή Ένωση, στα ειστάσια που αποφάσισαν οι πρόεδροι των Επιτροπών, οι διάσκεψη των Πρόεδρων, ε, τώρα το φθινόπωρο, οπότε έτσι θέλουμε να έχουμε τους διαδρομένους διαλόγους και με αυτόν τον πολιτικό διάλογο θέλουμε να ε, έχουμε μια συνένεση ευρεία όσον αφορά τις βασικές προτεραιότητες. Αυτό σημαίνει ότι μια που μπαίνουμε τώρα σε μια τέτοια περίοδο μεταβατική για τις εκλογές, οι πολίτες θα δουν ότι πραγματικά υπάρχει μια αίσθηση του ότι έχουμε μια κατεύθυνση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι θέλουμε να ολοκληρώσουμε την Τραπεζική Ένωση και ότι επίση θέλουμε να έχουμε ανάπτυξη και απασχόληση. Οπότε έτσι έτσι θέλουμε να τονίσουμε το ότι θα συνεχίσουμε αυτό μας το, τον ρυθμό, τόσο να ολοκληρώσουμε αυτές τις μεταρρυθμίσεις, ε, αυτές που κάναμε τα ε, πέντε τελευταία χρόνια, οπότε επίσης πέραν αυτών των πρωτοβουλειών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει εστιάσει την προσοχή της όσον αφορά την ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας, όσον αφορά κάποιες προτάσεις σημαντικές που ήδη έχουν τεθεί τραπέζης και θέλουμε να υπολογίζουμε την υποστήριξή σας για το έργο μας αυτό. Επίσης καλούμε τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν αυτό το οποίο έχουν ε, ε, συμφωνηθεί αμελητή. Επίση, θέλουμε να, έχουμε, να δούμε τι θα γίνει με το MFF, το πολιτέ πλαίσιο, και είναι πάρα πολύ σημαντικό ο ρόλο σα και έτσι καταφέραμε τη συμφωνία για τον νέο προπολογισμό που είναι καταλήτε για τι επενδύσει για, παντού. Οπότε και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Αυτά τα οποία ολοκληρώθηκαν για το MFF εχθέ και θα πρέπει να δούμε τώρα τα προγράμματα του MFF να ξεκινήσουν να τρέχουν όσο γίνεται συγκεκριμένα για να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα για του πολίτε και για τι επιχειρήσει επιχειρήσει κόντρα σε αυτή την κρίση, αγαπητοί κύριοι βουλευτέ, δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά και με δύσκολε συνεχεία, ούτω ώστε να δούμε το πώ θα μπορέσουμε να έχουμε την οικονομική ανάκαμψη και για να, να ξανακερδίσουμε την εμπιστοσύνη αγορών και Ευρωπαίων. Έχουμε κάποια καλά σημάδια σήμερα, αλλά δεν θα πρέπει να επαναπαυθούμε και αυτό, διότι θα πρέπει να κάνουμε παραπάνω βήματα χέρι-χέρι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ξεκινήσαμε το εξάμεινο το πρώτο για το 2014 τον προγραμματισμό την περασμένη εβδομάδα. Θέλουμε να είναι ισχυρή η κοινωνική πτυχή, αλλά πρόκειται για την πρώτη φορά για την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια αξιολόγηση όσον αφορά ε, τα σχέδια προπολογισμών ε, αυτό δημοσιοποιήθηκε την Παρασκευή, ούτως ώστε να δούμε πώ θα υπάρχει δημοκρατικό ε, έλεγχο. Οπότε θέλουμε να έχουμε ένα ενιαίο αποπτικό μηχανισμό, ε, ούτω ώστε να αλλάξει το τραπεζικό τοπίο και αυτό θα πρέπει να συνοδευτεί από τον ενιαίο μηχανισμό επίλυση ε, διαφορών. Το ίδιο αυτή την ανασυγκρότηση του κλάδου και τι άλλε συναφεί οδηγίε που θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλο τη κοινοβουλευτική θητεία. Να δούμε επίση πώ η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βοηθήσει εκείνου για του οποίου η ανασυγκρότηση ε, φαίνεται κάτι το μακρινό και όχι μια ρεαλιστική πιθανότητα. Θέλουμε να στηρίξουμε του νέου ε, άνεργου, αυτό για μα είναι προτεραιότητα. Επίση, να συνεχίσουμε να πιέζουμε τα κρατημέλη για να εφαρμόσουν ε, τι εγγύσει για την νεολαία για να αξιοποιήσουν τα κοινωνικά κονδύλια και να βοηθήσουν του νέου. Έχουμε ήδη έξι κρατημέλη που ξεκίνησαν αυτή την εφαρμογή συνεργασία μαζί μα. και επίση περιμένουμε και τα υπόλοιπα κρατημέλη να κάνω αυτό που πρέπει μέχρι το τέλος του έτους, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί το ότι αυτά τα 6 δις ευρώ για αυτή την πρωτοβουλία για την νεολαία θα απορροφηθούν όπως πρέπει επίσης όσον αφορά την κινητικότητα, όσον αφορά τη δικτύωση της δημόσιας υπηρεσίας, προσβασιμότητα σε χρηματοδότηση, όλα αυτά είναι προτεραιότητες και επίσης συμφωνήσαμε κάποιες αλλαγές όσον αφορά τους κανόνες της συνοχής και αυτό πρόκειται να προλυάνει το έδαφος για τις ΜΜΕ και το σχετικό χρηματοδοτικό μέσο. Επίσης παρακολουθούμε το τι θα γίνει για την πράσινη βίβλο, χρηματοδότηση, τόνωση της οικονομίας το 2014 Ακόμα έφραυστη υπόθεση η οικονομική ανασυγκρότηση, οπότε και εμεί θα πρέπει να διερευνήσουμε τι δυνατότητες της ενιαίας αγοράς να τις εκμεταλλευτούμε, έτσι να διαμορφώσουμε την ατζέντα μας και έτσι να είμαστε παντού ανταγωνιστικοί. Χρειάζεται η Ευρώπη μια βιομηχανική βάση ε, ισχυρή. Έχετε τις ε, προτάσεις σας για αυτές τις δύο, για τα δύο νομοθετήματα για την αγορά, για, για, τις, ε, για τις ηλεκτρονικές πληρωμές και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την ψηφιακή ενιαία αγορά. Ε, αυτό το, το θέλουν οι πολίτες. Επίσης η ενέργεια είναι μια μέρη ε, για όλους και γι' αυτό και εμείς θα πρέπει να συνεχίσουμε το έργο μας ώστε να μπορούμε να έχουμε μια αυθεντικά ενιαία αγορά για την ενέργεια. Επίσης θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει μακροπρόθεσμα για να δούμε τι θα γίνει με τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην ενέργεια θα πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε ένα πλαίσιο σαφές για κλιματικές και ενεργικές πολιτικές για μετά το 2020 εξότιμοι βουλευτές είμαστε μια κοινότητα αξιών οπότε ε, τώρα ελκύει την προσοχή μας η οικονομία αλλά δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς οι, οι ελευθερίες στηρίζουν την ευημερία, άρα αυτό όλα αυτά να τα περιφρουρήσουμε προς όφελος των πολιτών, θα πρέπει επίση να προστατεύσουμε τους πολίτες με προσαρμογή στι νέε απειλέ και προκλήσεις, συγκεκριμένη δράση χρειάζεται τους αμέσως μήνε για να δούμε τι θα γίνει με την προστασία των δεδομένων και να εξασφαλίσουμε το πώς οι επιχειρήσεις και οι πολίτες θα μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους με ασφάλεια. Επίσης, πρόκειται να προωθήσουμε αυτό που έχουμε σκεφτεί για το κράτος δικαίου και να συνεχιστεί ο προβληματισμό για το μέλλον τη Ευρώπη. Εχνούμε τον κοινό σκοπό να ολοκληρωθούν οι συνομιλίε για το καταστατικό και χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Γι' αυτό πριν έρθουν οι εκλογέ το 2014 θα συνεχίσουμε να περαμεινόμεθα των αξιών μα και των συμφωνών μα παντού σε όλο τον κόσμο. Θα πρέπει να καταδείξουμε ότι είμαστε κάτι το θετικό ε, παντού, να έχουμε ε, ανάπτυξη, να έχουμε ανθρωπιστική βοήθεια σε αυτούς που χρειάζονται, ε, να έχουν πολιτική γετνίαση, πολιτική διεύρυνση και να συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι μια όαση Ανάπτυξη Ειρηνικής. Ε, κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ, ήρθε η ώρα ούτω ώστε να, να, μπορέσουμε να κατευθύνουμε την ενέργειά μα, τι δυνάμει μα, ώστε να αξιοποιήσουμε όσο γίνεται περισσότερο τη σχετική νομοθεσία και όλε αυτέ τι σημαντικέ προτάσει να διεκπεριωθούν και να αρχίσουν να τρέχουν τα προγράμματα που σχετίζονται με το MFF. Οπότε και να συνεχιστεί η δική μα συνεργασία με εσά. Έχουμε κοινού στόχου και οι δύο θέλουμε το καλό για την Ευρώπη. Οπότε α συνεχίσουμε τη συνεργασία στο ίδιο πνεύμα, να κάνουμε ό,τι γίνεται περισσότερο και έτσι να δείξουμε στους πολίτες τι μπορεί να πετύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μια δηλαδή Ευρώπη που είναι ισχυρότερη, πιο ενωμένη και ανοιχτή σε όλο τον κόσμο. Και σας ε, ευχαριστώ και περιμένω πώς και πώς να τα συζητήσουμε αυτά. Ευχαριστώ εγώ κύριε Αντιπρόεδρε, λέει ο πρόεδρο και τώρα. Έχουμε τον πρώτο γύρο παρεμβάσεων από πλευρά των πολιτικών ομάδων. Πρώτα από και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Για δύο λεπτά και μισό έχει το λόγο ο κ. Σάγερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συνάδελφοι. Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα εργασία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2014, είναι πολύ σημαντικό να σεβαστεί τι αρχέ που ανέφερε και ο Επίτροπο. Δηλαδή, κατά πρώτον, το γεγονός ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε στις προτεραιότητες. Σε ό,τι αφορά το ΕΛΚ, οι προτεραιότητες αυτοί αφορούν λόγω χάρη τον εκβιομηχανισμό, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Εδώ σημαντική είναι επίσης η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, η πρόωθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η δημιουργία των απαραίτητων μέσων για την ε, Ευρωζώνη. Θα πρέπει τα στοιχεία αυτά να δοκιμάζονται κάθε φορά, διότι πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο εκπροσωπεί και προσφέρει προς τη θέμενη αξία στις εθνικές δράσεις. Οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν θα πρέπει να έχουν την αίσθηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παρεμβαίνει όπου ε, θα έπρεπε να αναζητούνται λύσεις σε τοπικό επίπεδο. Οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να έχουν την πεποίθηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται να συμπληρώσει τις εθνικές δράσεις και ότι εξυπηρετεί στην εξέβρεση λύσεων σε εθνικό επίπεδο. Αυτές λοιπόν οι δοκιμές, αυτά τα τεστ τη προστιθέμενης αξία πρέπει να γίνονται κάθε μία φορά ξεχωριστά. Κάτι άλλο που είναι επίση πολύ σημαντικό είναι ότι πρέπει να εξυπηρετήσουμε, να διευκολύνουμε τα κράτη-μέλη στο να βρίσκουν τι καλύτερε δυνατέ λύσει αλλά όχι χρησιμοποιώντας λύσεις πολυφορεμένες που δεν έχουν ε, δώσει αποτελέσματα. Είναι σαφές αυτό και για τους ε, κανονισμούς αλλά και για όλες τις δράσεις που προβλέπονται. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συνεισφέρει σε αυτή την προσπάθεια. Διότι και εμεί με τη σειρά μα θα πρέπει να έχουμε διεξαγάγει ήδη κάποια συμπεράσματα σε σχέση με το τι έχει γίνει στο παρελθόν. Το θέμα λοιπόν δεν είναι να παραμένουμε αδρανείς βλέποντας να αναζητούνται τοπικές λύσεις, αλλά να συνεισφέρουμε από τοπικές λύσεις δεν είναι δυνατές. Επίσης θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι αυτό είναι το έτος όπου το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αποδείξουν ότι η προστιθέμενη αξία που εκπορεύεται από το ευρωπαϊκό επίπεδο είναι κάτι απολύτως αναγκαίο και ότι δεν είναι κάτι επισκέπτο Ευχαριστούμε κύριε Σαγίδα. Δύο λεπτά τώρα και τους σοσιαλιστές. Έχει το λόγο ο κύριος Γερέρο Σολόμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να συνεχίσω πάνω σε αυτά που είπε στο τέλο τη ομιλία του Αντιπρόεδρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί πραγματικά θα πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί, ώστε να δείξουμε στου Ευρωπαίου στου αμέσω επόμενου μήνε ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε ή ε, στις προσδοκίες τους και τα όσα χρειάζονται. Δεν θέλω ε, εμείς να, ε, να, είμαστε σε κάποιο είδου αναπηρία το επόμενο εξάμεινο. Θέλουμε την άλλη μεριά να κάνουμε ό,τι γίνεται, ό,τι είναι δυνατόν, τόσο ώστε να ανταποκριθούμε σε όσα χρειάζονται και γι' αυτό θέλουμε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε ε, την κατάρτιση κάποια λίστας με προτεραιότητες. Πρώτα απ' όλα να δούμε το πώς θα έχουμε ποιοτική απασχόληση, πώς θα προστατεύσουμε τους εργαζόμενους, όλους τους εργαζόμενους, αλλά ιδίω θέλουμε να δούμε τι θα γίνει με εκείνους που έχουν αποσπαστεί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αυτή τη στιγμή τώρα τίθενται ένα αμφιβόλο και εγκινδύνω τα δικαιώματά τους σε μια σειρά ε, ε, χώρων. Πρώτα-πρώτα όμως θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε την ανεργία των νέων, γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή 15 χώρες που έχουν ανεργία στους νέους 20 με 30% και 6 αυτές οι χώρες έχουν πάνω από 3%, 4 πάνω από 40%, 2 χώρες πάνω από 50%. Πρόκειται επίσης για 6 χώρες μόνο οι οποίες έχουν εγκρίνει τα προγράμματα για την εγγύηση για την νεολαία. Θα πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε ε, ε, κατά των ε, ανισοτήτων και κατά της περιφερειακής εδαφικής συνοχής να δούμε τι θα γίνει με την μακρορεσιμότητα να δούμε πώς θα επιβάλλουμε κάποιες και τι θα κάνουμε τις χώρες εκείνες που χρειάζονται ε, ε, τους πόρους, η κυρώση δεν ήταν λάθος, ε, πάντως θα πρέπει να δούμε το τι θα γίνει με τη συρρήγνωση των πόρων του κοινωνικού ταμείου. Αυτό έγινε τώρα σε συγκυρία κρίση. αυτό είναι λάθος. Αυτό είναι τελείω λάθος κατεύθυνση. Πρέπει το 25% του συνόλου να το προσθέσουμε τόσο ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη σημερινή ε, κοινωνική πολιτική αυτή που ασκεί τώρα το ΕΚΤΑΦ. Να μην συγγνώμη αυτή την πολιτική. Ακριβώ τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να γίνει αυτό, γιατί το αυτή πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την χωρί προηγούμενο κρίση. Ο πρώτο Ενρίκη, ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα. Του φιλελευθέρου. Ο φίλο Άντριου Ντάφη, το λόγο. Η ομάδα των Ελευθέρων, κύριε Πρόεδρε, χαιρετίζει αυτό το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτές τις ε, λιτές προτεραιότητες σε σχέση με την καινούργια εντολή και επίσης θα πρέπει να πούμε γενικώ ότι αυτή η διαδικασία για την κατάρτιση του προγράμματος εργασίας είναι κάτι το οποίο αποδίδει καρπούς και έπιασε όσον αφορά τη συνεργασία Κοινοβουλίου και Επιτροπής. Αυτό πάντως στο οποίο πάσχει είναι το ότι δεν συνέπλευσε το Συμβούλιο το έχουμε ένα κοινό πρόγραμμα εργασίας και για τα τριθεσμικά όργανα τελικά καταλήξαμε να έχουμε αυτού του είδους τα προγράμματα προεδρίας που είναι σε στυλ Τρόικα θεωρούμε ότι αυτό δεν βοηθάει δεν είναι ε, λογικά συνεπές, δεν διακρίνεται από λογική συνοχή, άρα ήρθε η ώρα να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας από πλευράς νομοθετικής Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να αναλάβει τα ενία προς τη σωστή κατεύθυνση και να μπορέσει να διαχειριστεί τα θέματα τα οποία προκύπτουν από τα συνήθεια τακτικά συμβούλια. Θα έχουμε ένα νέο κοινοβούλιο, θα έχουμε μια νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή που πρόκειται να προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν την εμπλοκή του Συμβουλίου στη διαμόρφωση των προγραμμάτων εργασία ή στο μέλλον. Άντρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. και τώρα για του πρασίνου. Ένα λεπτό. Γιάννη Ζαντό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, αγαπητοί συνάδελφοι, οι διαπραγματεύσει για την συνθήκη των ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών με τις ΗΠΑ είναι κάτι που θα απασχολήσει πάρα πολύ σοβαρά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρετε ότι μιλάμε για κοινωνικέ επιλογέ που είναι αντικείμενο διαπραγματεύσεων, για τι κοινωνικέ υπηρεσίε, την προστασία των καταναλωτών, για τα δικαιώματα των επενδυτών, για του γενετικώ τροποποιημένου οργανισμού, για το βοδινό με ορμόνε, για την προστασία μα γενικώ. Οι διαπραγματεύσει όμω αυτή γίνεται με πλήρη αδιαφάνεια σε σχέση με τα όσα μπορούν να παρακολουθήσουν οι Ευρωπαίοι πολίτε. Μιλάτε για δημοκρατία, για κοινότητα αξιών. Πώ η στάση και η συμπεριφορά του Συμβουλίου και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που απαγορεύουν αυτή τη στιγμή στου Ευρωπαίου πολίτε να έχουν πρόσβαση ακόμα και μόνο στην απλή διαπραγματευτική εντολή, πώ αυτό ενισχύει τη δημοκρατία στην Ευρώπη. Ξέρετε ότι ενισχύει την αντίληψη των Ευρωπαίων πολιτών ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση απλώ εξυπηρετεί τι πολυεθνικέ εταιρείε. Και αυτό ει βάρο των συμφερόντων των ίδιων των πολιτών. Η ομάδα των Πρασίνων λοιπόν σα ζητά ρητός να υπάρχουν διαπραγματεύσεις πλήρω διαφανείς και οι Ευρωπαίοι πολίτες να γνωρίζουν πώ ακριβώς διαπραγματεύεστε το μέλλον της κοινωνίας τους. για 1,5 ε, Ευχαριστώ κυρίε και κύριοι. Η πρώτη αρμοδιότητα και το πρώτο καθήκον οποιασδήποτε Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η εξέταση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας από την πλευρά της ανταγωνιστικότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα φαίνεται να είναι υπεύθυνη για την μείωση ε, της οικονομικής δραστηριότητας ε, των Ευρωπαίων πολιτών. Έτσι το αντιλαμβάνονται. Ε, θα πρέπει να μειωθεί όμως το διοικητικό άχθος, ο γραφειοκρατικός φόρτος που έχει επιβληθεί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να υπάρξει απελευθέρωση της αγοράς των υπηρεσιών και της ψηφιακής αγοράς. Χρειάζονται νέα κέρδη και όλο ένα προτείνουμε νέους κανονισμούς. Οι κανονισμοί αυτοί πρέπει να εξετάζονται από τη σκοπιά ε, του αντικτύπου που θα έχουν στην ανταγωνιστικότητα. Θα πρέπει να έχουμε λίγους μεν κανονισμούς αλλά που να είναι ε, αξιοποιήσιμη από τους επενδυτές. Ιδίω ό,τι αφορά την Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κοινή αγορά σήμερα είναι το μόνο εργαλείο που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε την κρίση και θα πρέπει να το επανεπινοήσουμε. Ευχαριστούμε κύριε Σιμάνσκι. Και τώρα εκ μέρου ε, της Ευρώπης για τη Δημοκρατία και την Ελευθερία, 1,5 λεπτό για τον κύριο Πάξας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, του χρόνου η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κληθεί να αντιμετωπίσει μια σειρά προκλήσεων. Οι βασικότερες είναι η ε, ανάκαμψη της οικονομίας με αηφορία και μείωση της ανεργίας. Υποστηρίζω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η πρώτη προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η οικονομική ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασίας με ιδιαίτερη εστίαση στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Καθώς επίσης και τη διευκόλυνση ε, στην πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα πρότεινα να είμαστε πιο ε, συγκεκριμένοι στη δράση μας. Τι εννοώ. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση αποπειράται να ε, ορίσει το μέγεθος της μπανάνας, του αυγού ή του αγγουριού. Έχει νόημα αυτό τώρα να λέμε πιο ε, είναι το μέγεθος και τα μέτρα και τα σταθμά. Τώρα θέλουμε λέει να έχουμε ένα ενιαίο κατώτατο μισθό. Εδώ φωνάζουμε δεξιά και αριστερά ότι πρέπει να ενισχυθεί η ενιαία αγορά. Μα δεν θα είναι ποτέ ισχυρή η ενιαία αγορά, ενώ το 1 πέμπτο των Ευρωπαίων ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Εγώ πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ψάξει νέους τρόπους και να αναζητήσει ευκαιρίες και δυνατότητες ενίσχυσης της εργασίας των νέων στα κράτη-μέλη. Θα μπορούσαμε να επιδοτούμε εργοδότες ενδεχομένω να μειώσουμε ε, τη φορολόγηση της εργασίας ή εκεί να έχουμε ομοιόμορφα μέτρα ε, να μειώσουμε ας πούμε, τη φορολογία για εκείνους που απασχολούν νέου μέχρι ηλικία 30 ετών. Ευχαριστώ. Τελευταίο συνάδελφος που θα μιλήσει εξ ονόματος των μη εγγεγραμμένων σε αυτή τη συζήτηση για 1,5 λεπτό είναι ο κύριος Μποργέζιο. Κύριε Πρόεδρε, μετά τη Λαμπεντούζα πολλά μεγάλα λόγια ακούστηκαν για την μετανάστευση. Κανένα όμω πεπραγμένο. Ε, ακόμα και το πρόγραμμα για το 2014 περιλαμβάνει πολύ λίγα στοιχεία. Εδώ χρειάζεται μια συγκεκριμένη ε, ε, άμεση αντίδραση στρατηγική για να αντιμετωπιστούν αμέσω αυτέ οι ροέ που προκαλούν τραγωδίε όπω αυτή τη Λαμπεντούζα. Μιλάμε για τον Δημοσιονομικό Κανονισμό και την Τραπεζική Ένωση. Μια ερώτηση. Τι περιμένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πώ συσχετίζει και πώ έρχεται εδώ και μιλάει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το τι συμβαίνει με τις, αγνοεί τι συμβαίνει με τις γερμανικές τράπεζες. Είναι γνωστό σε όλο τον κλάδο ότι υπάρχουν τεράστια ποσά παραγόγων που αποθηκεύονται στις γερμανικές τράπεζες και καταλήγουν σε φορολογικούς παραδείσους. εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και αυτά διασώζονται με κρατικές βοήθειες. Ιδίως στον ε, τομέα της γερμανικής τραπεζικής δραστηριότητας. Εδώ λοιπόν η αντιμετώπιση των φορολογικών παραδείσων είναι μια κατεπίγουσα προτεραιότητα για να υπάρξει μια απόκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να είμαστε. Και θέλω εδώ μια απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα. Λέτε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Τι γίνεται με τι μεταφορέ για του Ευρωπαϊκού πολίτε. Τι γίνεται με την κατακαμένη την Σαρδινία η οποία πλημμυρίζει δεν υπάρχουν δρόμοι για να πάνε οι βοήθειε εκεί που πρέπει. Είναι λοιπόν τελείως φάλτσα τα λόγια που ακούγονται και η Σαρδινία από το Ιταλικό κράτος αντιμετωπίζεται ως απικία και προφανώς και ε, επιζητά την ανεξαρτησία της και την αυτονομία της. Πρέπει να μην ξεχνάμε την πραγματικότητα κάποιων περιφερειών που κάποια κράτη-μέλη τις αντιμετωπίζουν λες και ήταν απικίες. Η Σαρδινία αυτή τη στιγμή χρειάζεται βοήθεια και αλληλεγγύη, αλλά χειροπιαστή, διότι σκεφτείτε σε τι συνθήκε την εγκατέλειψαν. Ε, για την τραγωδία αυτή είναι υπεύθυνοι όσοι ε, έχουν συγκαλυφθεί και από πολιτική σκοπιά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Συνάδελφε, τελείωσε ο χρόνος σας. Για να κλείσει η συζήτηση θα ακούσουμε και πάλι τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα απαντήσει στα λεγόμενα των βουλευτών. Κύριε έχετε το λόγο, παρακαλώ. Thank you very much, uh, Mr. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές οι οποίοι θεώρησαν ότι είναι πάρα πολύ εύστοχο, ευσύνοπτο το πρόγραμμά μας 2014 και θα πρέπει να σας ε, βεβαιώσω ότι δεν ήταν καθόλου εύκολη η κατάρτιση του πίνακα των προτεραιοτήτων, γιατί έχουμε τόσε εκατοντάδε ε, προτάσεις, αλλά εμεί θα έπρεπε να ξεκαθαρίσουμε σαφώς την εσωτερικότητα περίπου 26, οπότε είδατε ότι εκεί είναι καλύτερα να εστιάσουμε το έργο μας για όσο απομένει ε, για αυτήν την ε, νομοθετική κοινοβουλευτική περίοδο, για όλε αυτές τι προτάσει που θα μα οδηγήσουν στην όσο γίνεται περισσότερη προστιθέμενη αξία για την Ένωση και που να συμβάλλουν όσο γίνεται περισσότερο στην δημιουργία απασχόληση και οικονομική ανάπτυξη. Όπω μπορείτε να διαπιστώσετε από τα παραρτήματα, για πρώτη φορά έχουμε εδώ. Πρώτη φορά εδώ πέρα μνημονεύουμε το REFIT, τόσο ώστε να μπορέσουμε να έχουμε λιγότερη γραφειοκρατία. Επίσης στις προτεραιότητες βλέπετε ε, κάποια σχέδια οδηγιών και κανονισμών με τα οποία ελπίζουμε ότι θα πετύχουμε αυτό το οποίο θέλουμε για την επόμενη περίοδο. Επίσης, ε, όσον αφορά το όσο είπε ο κύριος Ντάφ, μας είπε ότι χρειάζεται καλύτερο προγραμματισμός στο μέλλον. Αυτά που είπε είναι σύμφωνα με αυτά τα οποία συζητήσαμε χτες και τα οποία συζητήσαμε στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων. Πρέπει να κάνουμε καλύτερη εφαρμογή, υλοποίηση, να κάνουμε καλύτερο προγραμματισμό, να ε, συντονίζουμε ε, το έργο μας με τα όσα γίνονται στις ομάδες εργασίας του Συμβουλίου και έτσι επομένως όλοι χέρι-χέρι παράλληλα να προωθούμε τις προτεραιότητές μας. Πολύ υπουργοί αναφέρθηκαν στο Συμβούλιο στο ότι μετά τι επόμενε εκλογέ θα πρέπει γύρω από ένα τραπέζι να κάνουν τρία θεσμικά οργανά και να εξετάσουν ε, την ισχύουσα ε, συμφωνία πλαίσιο, αυτή που συνυπογράψαμε και έτσι να δούμε ε, πώ θα συμφωνήσουμε εμεί με το Συμβούλιο για να μπορέσουμε έτσι να έχουμε περισσότερο και καλύτερο προγραμματισμό στο μέλλον. Σα διαβεβαιώ, από δική μα πλευρά είναι πολύ σημαντικό να ακολουθούμε την κοινοτική μέθοδο και επίσης να τηρείται το προνόμιο ε, της πρωτοβουλίας που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, μας είπατε για ε, ε, αυτό το που θα κάνουμε τον Ιανουάριο θα εκδώσουμε μια ανακοίνωση όπως τα είπατε για να αναλύσουμε το τι θα κάνουμε με τις ενεργειακές τιμές γιατί είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας και για αυτό και θα, αυτές οι ανακοινώσεις θα δημοσιευθούν ταυτόχρονος και θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Πολύ σωστά είπε ο κύριος Γκερέρο ότι το βασικό μας πρόβλημα σήμερα είναι η ανεργία. Ξέρουμε ότι για να αντιμετωπιστεί σωστά χρειάζεται ανάπτυξη καλύτερη, σταθερότερη και θα πρέπει επίσης να μην ξεχνούμε το ότι συνήθως ε, υστερούμε όσον αφορά την απασχόληση έξι μήνες με ένα χρόνο σε σχέση με τους ρυθμούς που τρέχει η ανάπτυξη. Οπότε θα πρέπει να δημιουργήσουμε γίνεται και τα μέλη και να προχωρήσουν στον αφορά αυτού του είδους τα προγράμματα εγγύησης για την νεολαία γιατί ιδίω των νέων η ανεργία βρίσκεται πάρα πολύ ψηλά. Άρα θα πρέπει από τον Ιανουάριο του επόμενου έτους να αξιοποιηθούν οι κοινοτικοί πόροι. Στον κύριο Πάξα θέλω να πω ότι θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την φορολόγηση εργασία. Πιέζουμε, απευθύνουμε συστάσει στα κράτη-μέλη, το συμβουλεύουμε τα κράτη-μέλη να εγκαταλείψουν το μοντέλο της υπερβολικής ε, φορολόγησης ε, της ε, εργασίας και να έχουν μια φορολογία φιλική στην ανάπτυξη, ούτως ώστε να μην ε, αποθαρρύνεται η κινητικότητα, η δημιουργία εργασίας, γιατί θέλουμε τη δημιουργία τη εργασία. Θέλουμε να υπάρχει προσαρμογή της φορολογικής πολιτικής ε, με την, και ε, στην πολιτική απασχόληση. Επίση, ευχαριστούμε που τονίσατε το πόσο σημαντικό είναι να αντιμετωπίσουμε τη γραφειοκρατία, πότε είναι σημαντικό να νομοθετήσουμε σχετικά και να καταλήξουμε έτσι στο να έχουμε προσθεμενή αξία. Τα είπαμε χτε με τους υπουργούς την ώρα που και εδώ τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Πρέπει να είναι κοινή η προσπάθεια, πρέπει να κάνουν τέτοιες προσπάθειες, θα πρέπει να μειωθεί η γραφειοκρατία. Αλλά βέβαια η σχετική πρόταση θα πρέπει οι συνομοθέτες να την εγκρίνουν. Αλλά θα πρέπει βέβαια να μεταφερθεί όπως πρέπει στα κράτη-μέλη τα οποία ε, να προσέξουν, να μην περιπλέξουν την εφαρμογή ε, με επικαλύψεις γιατί έτσι αυξάνεται η γραφειοκρατία χρειάζεται κόπος. Θα έχουμε τις εκθέσεις, θα έχουμε τους πίνακες επιδόσεων, έτσι θα παρακολουθούμε το τι κάνουν τα κράτη-μέλη, πώς τα πάνε, όσον αφορά τις προσπάθειες που καταβάλουν για να μειωθεί αυτή η γραφειοκρατία. Και σε εθνικό επίπεδο. Οπότε γι' αυτό και θεωρούμε ότι τελικά από όλα αυτά θα βγει μια κατάσταση υγιούς, ανταγωνισμού, οπότε θα είμαστε σε θέση να κάνουμε έναν ε, θετικό απολογισμό σε ένα χρόνο ω Βοργέζιο μας είπε για την τραγωδία της Λαμπεντούζα. Τον ενημερώνω ότι η Task Force για τη Μεσόγειο δουλεύει ακάματα για αυτή την έκθεση που θα καταρτήσουν τόσο ώστε να διατυπώσουν κάποιες προτάσεις. Θα τα συζητήσουμε εδώ στο Κοινοβούλιο αλλά και στα συναρμόδια συμβούλια. Για το TTIP έχουμε τις ε, διαπραγματεύσεις με ε, τις Ηνωμένε Πολιτείε. Είπαμε ότι ετησίως διακυβεύονται 190 ε, δις γιατί θα πρέπει να δούμε για αυτή την εμπορική συμφωνία τι θα γίνουν τα νέα πρότυπα, με τις νέες τεχνολογίες. Γι' αυτό είναι σημαντικό να προστατεύσουμε τις προτεραιότητές μας, να διαπραγματευόμαστε με φιλοδοξία. Ε, αυτό και κάνουμε, γιατί ξέρουμε ότι αυτό είναι ό,τι καλύτερο χρειάζονται οι Ευρωπαίοι και οι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει. Ευχαριστώ και πάλι, κύριε Διπρόεδρε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θα ήθελα να κλείσω τη συζήτηση χωρί να τονίσω πόσο ευχάριστο ήταν πάντα ε, συνεργαζόμαστε και θα μας λείψετε. Αναφερθήκατε στις επόμενες εκλογές και γνωρίζετε όλοι ότι κάθε φορά που υπάρχουν εκλογές πάντα κάποιος υπουργό έρχεται στο Κοινοβούλιο ε, ή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, και γίνονται επίτροποι οι βουλευτές και ελπίζω να μάθουν πολλά οι υπουργοί ε, αυτοί και με τον ίδιο ενθουσιασμό ε, να αγωνιστούν για την ε, κοινοτική μέθοδο, με το ίδιο σθένος που είχαν αγωνιστεί για τη διακυβερνητική συνεργασία όταν ήταν υπουργοί. Σας ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση αυτή. Α, ζητώ συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος. Στη συζήτηση αυτή δυστυχώς δεν υπάρχει διαδικασία ΚΑΤΣΙΑ. Έχει τελειώσει. Για διαδικαστικό θέλετε κύριε Ζαντό, παρακαλώ, αλλά πάρα πολύ σύντομα σας παρακαλώ. Ναι, είναι διαδικαστικό κύριε Πρόεδρε, διότι ο κύριος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σκηνοθετεί και ομιλεί για τη συνεργασία με το Κοινοβούλιο και εγώ το ρώτησα κάτι για τη διαφάνεια των διαπραγματεύσεων και δεν μου απάντησε. Ε, Θέλω εδώ όταν έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντά και ε, στο Ευρωπαϊκά Δημοκρατικά εκλεγμένο σώμα των βουλευτών. Κοιτάξτε, λέει ο Πρόεδρος, απάντησε ως ενόμιζε ε, ο Επίτροπος και μπορεί ο καθένας έχει το δικαίωμα να μένει ικανοποιημένος ή δυσαρεστημένος από την απάντηση. Λοιπόν, να σας δώσω τώρα κάποιες λεπτομέρειες για τη διαδικασία. Ε, θα διακόψουμε για λίγο και επίσημα μέχρι τις 12.30 δεν επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση ε, που θα επαναληφθεί στις 12.30 για την ψηφοφορία. Αλλά στις 12 ελπίζω να είστε όλοι παρόντες και να είμαστε γιατί ε, έχουμε την απονομή του βραβείου Ζαχάροφ. Ορίστε, τι θέλετε, και εσείς διαδικαστικό έχετε, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Την Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μάλλον κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να σας πω ε, ότι ε, γιορτάζουμε την επέτειο ε, της μάχης του Βούκοβαρ και θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε Κροάτες ε, παλεμάχους ε, στο θεωρείο και θα ήθελα να τους καλωσορίσουμε. Γνωρίζετε αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι ότι έχω επανειλημμένα μεταβεί στο Βούκοβαρ και όταν εορτάσαμε ε, το σπίτι των εργατών και την ανοικοδόμηση του θαυμάσιου αυτού κτηρίου. Ε, και πραγματικά είμαι πολύ προσιλωμένο στα θέματα αυτά και με συγκινεί και με χαροποιεί το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ε, προεδρεύω παρουσία των διακεκριμένων μας προσκεκλημένων. Λοιπόν, διακόπτεται εδώ η συνεδρίαση μέχρι τις 12 και 12.30 αντίστοιχα για τις δύο υποθέσεις που έχουμε ακόμα στη σημερινή πρωινή συνεδρίαση. Ευχαριστώ